Chers collègues, la séance est reprise. Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε. Ελπίζω να έρθει η Ιζαμπέλ αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε. Διότι σύμφωνα με τη μέσα διάταξη έχουμε πολλά να πούμε. Και κυρίως το πρώτο, προετοιμασία το συμβαστικών προτάσιο για τις αυριανές ψηφοφορίες για την έκθεση πρωτοβουλίας για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 και την έκθεση πρωτοβουλίας για τους νέους ίδιους πόρους. Οι συνεισηγητές θα παρουσιάσουν τις συμβαστικές προτάσεις και τις κύριες συστάσεις τους εν ώψη της αυριανής ψηφοφορίας. Λοιπόν, θα ξεκινούσαμε με το πολιτές πλαίσιο, αλλά επειδή λείπει η Ζαμπέλτομα Τόμα, μήπως να αρχίσουμε με τους νέους ίδιους πόρους. Γιατί Ζεράρ Ντεπρέ και Λεβαντόφσκι είναι παρόντες. Δεν θα ξανακάνουμε τη συζήτηση. Όχι. Θα συζητήσουμε την επίτευξη συμβαστικών προτάσεων και θα ακούσουμε τις απόψεις των μεν και των δε. Ποιος θέλει πρώτο το λόγο, ο κύριος Ντεπρέ ή ο κύριος ε, Λεβαντόφσκι. Και μετά στους Κιώδης, επί των προτάσεων, συμβιβασμού, που θα ψηφιστούν αύριο πρωί. Ο κύριος Λεβαντόφσκι. Κανείς δεν περίμενε να είναι εύκολη αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ τους σκιώδες και τους συνεργάτες μας για τη συνεργασία. Θέλουμε να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο πριν τοποθετηθεί ο Έτιγκερ και να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να επιδείξει θάρρος για το θέμα των ε, ιδίων πόρων. Έχουν υποβληθεί την τροπολογίες. Οι περισσότερες είναι υπέρ ε, των ε, ίδιων πόρων. Οι περισσότερες θέλουν να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα για τα έσοδα της Ένωσης. Πολύ καλή συνεργασία. Κατέληξε σε 34 συμβιβαστικές. Βεβαίως δεν μας εκπλήσει το ότι συμφωνήσαμε επί των αρχών για την τροποποίηση των εσόδων και για την αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήματος. Τώρα δεν θα συζητήσω μία-μία τις τροπολογίες. Αυτό που είναι σημαντικό, όπως λέει η Συμβαστική Τροπολογία 1, είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν θα αποδεχθεί το ΠΔΠ αν δεν υπάρχει ένα σαφέ πλαίσιο για τους ίδιους πόρους. Και αν δεν ε, δηλωθεί σαφώς, όπως λέει και η Συμβαστική 3, ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την έννοια του καθαρού συνεισφορέα, καθαρού αποδέκτη και πρέπει να χρηματοδοτηθεί το κενό που θα προκύψει από τον Brexit. Αλλά ε, δεν μας εκπλήσει επίσης το ότι ήταν πιο δύσκολο να συμφωνηθούν ορισμένα άλλα θέματα, αλλά και εδώ έχουμε κάποιες συμβαστικές. Δηλαδή, ποιοι μπορεί να είναι οι νέοι ήδη οι πόροι. Ε, πάνω κάτω λέμε και αυτά που λέει και το προπαρασκευαστικό κείμενο της Κομισιόν για την αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου. Γιατί εάν δεν αλλάξει η ημερήσια διάταξη για την αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου, θα ικανοποιηθεί ο στόχος του Κοινοβουλίου να υπάρξει τελική συμφωνία πριν από τις εκλογές. Ως συνεισηγητής, το πιο δύσκολο ήταν ότι οι ίδιοι πόροι θα πρέπει να βοηθήσουν την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ε, πορεία προς την οικονομία χαμηλού άνθρακα. Εδώ συμφωνούμε με τους πρασίνους. Και θέλαμε να υπάρχει μια τροπολογία επί, την οποία να επί της οποίας να συμφωνούν όλοι. Έχουμε μια σειρά από ενδεχόμενους νέους ίδιους πόρους που θα μας βοηθούσαν να περάσουμε σε μια οικονομία χαμηλού διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά Θέλουμε επίση να καταργηθούν και όλες οι εκπτώσεις. Γιατί δεν έχουμε μόνο τη Βρετανική έκπτωση. Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτές τις διορθώσεις και τις εκπτώσεις, γιατί είναι πολύ περίπλοκο αυτό το σύστημα, όπως λειτουργεί σήμερα, και αν χρειαστούν κάποιες αντισταθμίσεις, δεν θα πρέπει να γίνουν στην πλευρά των εσόδων, αλλά μέσω ειδικών προγραμμάτων δαπανών. Αυτή είναι η συμφωνηθής αρχή για την εντεχόμενη ε, αντιστάθμιση για την κατάργηση κάποιων εκπτώσεων. Γιατί αυτό θα επιβαρύνει κάποια κράτη-μέλη. Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες ε, αρχές επί τις οποίες συμφωνήσαμε. Επί... Ναι. και ο κύριος Λαμασούρ που έκανε τόσο πολλά στο παρελθόν πρότεινε να υπάρξουν για σύντομο χρονικό διάστημα κατά αποκοπήν ποσά. Γιατί δεν είναι εύκολο να ε, καταργήσουμε όλες τις ε, διορθώσεις. Αλλά η αρχή μας είναι οι αντισταθμίσεις, οι αποζημιώσεις να είναι όχι μέσω διορθώσεων στην πλευρά των εσόδων, αλλά μέσω ειδικών προγραμμάτων δαπανών. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Αυτά συμφωνήσαμε με τον Ζεγά, ε, με τον οποίο ε, είμαστε δύο συγκεκριτές μια φωνή. Και... Ευχαριστώ. Θα ακούσετε μια άλλη φωνή για τα ίδια θέματα. Ε, είμαστε όμως ένα μέτωπο. Δύο άνθρωποι, ένα μέτωπο. Γι' αυτό θα είμαι συντομότατος. Ευχαριστώ τον συνεισηγητή μου, γιατί δουλέψαμε με αγαστή συνεργασία. Ε, γνώρισαμε κάποιες πιο έντονες στιγμές, αλλά τελικά και οι δύο, και χάρη στους δύο και σε απόψεις και των δύο, ε, εξασφαλίζουμε αυτήν την ισορροπία. Για να μην το ξεχάσω, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες της γραμματείας της ομάδας, το ξέχασα σήμερα το πρωί, για την αμεροληψία τους και την λεπτότητά τους. Μερικές φορές ε, τους θαύμασα. Ε, θαύμασα τη συμπεριφορά τους και τους χειρισμούς τους και το πώς στάθηκαν απέναντί μας. Λοιπόν, τώρα. Κάνω έκκληση ε, στους όλους τους βουλευτές να ξαναθυμηθούμε αυτή την βασική αρχή. Οι νέοι διπόροι να είναι η ε, αναπόσπαστο τμήμα της ε, έκθεσης για το που πουδουπού. Δηλαδή, να μην συμφωνήσουμε το επόμενο πουδουπού αν δεν έχουμε και ένα κεφάλαιο για τους ίδιους πόρους. Τελεία. Κατά τα άλλα, δεν δυσκολευτήκαμε γιατί είχαμε την έκθεση της ομάδας Μόντι και τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε τα παίρνουμε από τις προτάσεις που είχε κάνει η ομάδα Μόντι. Προσθέσαμε και ένα στοιχείο βέβαια σε ό,τι αφορά το εξής. που αφορά την ε, παγιοποίηση του εταιρικού φόρου. Ε, περιμένουμε δηλαδή από τις, ε, εταιρικές, από τις ψηφιακές εταιρείες να συνεισφέρουν κι αυτές. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες που θέλουν να εξελιχθεί καλά η Ευρώπη, νομίζω ότι μπορούν να συμφωνήσουν ε, με τις αδρές γραμμές αυτής της έκθεσης. Βλέπετε ποια είναι η φιλοδοξία, βλέπετε το ρεαλισμό. Αυτά. Ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές που μας υπέβαλαν μια πλήρη έκθεση. Και ευχαριστούμε και αυτήν την αναφορά που έκανα στην ομάδα Μόντι, που ήταν μια ομάδα η οποία αποτελούνται από εκπροσώπου των τριών θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Και επομένως δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε για την αποφασιστικότητα του Συμβουλίου να υλοποιήσει τους, αυτό το κεφάλαιο των νέων ε, ιδιών πόρων. Επίσης, για αυτό τον άξονα για τον οποίο λέγατε, ε, έχετε μερικές χώρες που έχουν ε, πολλές, πολλούς, πολλές εταιρείες και άρα ε, πολλούς εταιρικούς φόρους. και από την άλλη έχετε χώρες οι οποίες δεν βάζουν τόσους φόρους στις εταιρείες. Ε, πρέπει να λύσουμε αυτήν την διαφορά. Μερικές ε, χώρες φορολογούν πολύ τα, τα, εταιρικά κέρδη. Αλλά σε άλλες χώρες που έχουμε περισσότερες, μάλλον λιγότερες εταιρείε, πολλές όμως πρόσωποπαγεί εταιρείε και άρα ε, περισσότερους τέτοιου φόρους, θα πρέπει να, κάπως να παντρέψουμε αυτές τις διαφορές. Τώρα θα δώσω το λόγο στου σκιώδεις εισηγητέ. Ο, Φερ... ο κύριος Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες είναι ο πρώτος ε, σκιώδης εισηγητής. εκφράστηκε ήδη μέσω του εισηγητή. Άρα δεν πρέπει να ακούσουμε τον Χωσέ Μανουέλ. Φοντανιέλε, διότι θα μιλήσει εξ ονόματος των σοσιαλιστών που δεν ε, εκπροσωπείται στην, ε, στο δίδυμο Λεβαντόφσκι Ντεπρέ. Η ομάδα των σοσιαλιστών δεν εκπροσωπείται σε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν, αυτή την τελευταία μας συζήτηση θα ήθελα να την ξεκινήσω ευχαριστώντας τους δύο συνεισηγητές που έκαναν μια δουλειά πλήρη όπου βρίσκουμε πολλές από τις δικές μας πολιτικές διεκδικήσεις τουλάχιστον της ομάδας που εγώ εκπροσωπώ σε αυτή τη συζήτηση. Πολλά επίσης από τα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Στο εσωτερικό μιας Ευρώπης που θα πρέπει να είναι πιο ομοσπονδιακή, πιο ικανή να ανεφοδιαστεί από μόνη της, αν θέλετε, οικονομικά. Επίσης, ο κ. Ντεπρέ ανέφερε την ομάδα Μόντι. Όταν ε, συναντήσαμε για πρώτη φορά την ομάδα Μόντι, την ομάδα υψηλού επίπεδου Μόντι και τον πρόεδρό τη, τον κύριο Μόντι, στην Επιτροπή μας, ο πρόεδρος Μόντι μας ε, παρουσίασε μια εκθεσούλα ε, που την έλεγε η γκρίζα έκθεση. Γιατί ήταν απλώς κάποια, ήταν ένα σκαρίφημα ας πούμε, δεν είχε πολύ ψωμί μέσα, πολύ... ήταν ένα σκελετός ας πούμε. Τώρα όμως βλέπετε ότι είναι μια έκθεση πολύ πιο πλούσια. Κάτι παραπάνω από αυτήν την γκρίζα έκθεση που ήταν στην αρχή. Η τελική έκθεση ο ομάδας Μόντι. Τώρα, αυτά ευχαριστώντας τους δύο συνεισηγητές για τη δουλειά που κάνανε. Τώρα, κάτι που δεν υπάρχει ακόμα και που δεν ακούστηκε στην έκθεση. Παρά την τεράστια δουλειά που, που έγινε, φτάνουμε λαχανιασμένοι, ας πούμε, στην γραμμή άφηξης. Ακόμα δουλεύουμε, ακόμα τελευταία στιγμή ψάχνουμε το κείμενο, βάζουμε, κόβουμε, ράβουμε κτλ. Είμαστε στο τσακ να φτάσουμε, να ολοκληρώσουμε ε, την έκθεση αυτή, αλλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, όχι στα μεγάλα θέματα, ευτυχώς αλλά σε κάποιες λεπτομέρειες, που όμως έχουν μια πολιτική σημασία για διάφορους από εμά, πούμε, για, τον α, το τάδε θέμα, για τον β κάποιο άλλο θέμα. Ελπίζω, για να είμαι σίγουρο, ότι μέχρι να τελειώσουμε τη σημερινή συζήτηση, τη γενική συζήτηση, θα καταφέρουμε να βρούμε και συμβιβαστικέ λύσει ακόμα καλύτερε. Και έτσι αύριο θα είμαστε πολύ χαλαροί και θα έχουμε όλοι αυτό που επιθυμούμε. Δηλαδή, μία καλή ψήφο, πλατιά, πλατιά πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας αυτής των ε, συναδέλφων Λεβαντόφσκι και Ντεπρέ για τους ε, ίδιους πόρους και για την έκθεση για το Πουδουπού, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον ε, Τωμά Ολμπριχτ, που θα πρέπει να εγκριθούν αύριο το πρωί πριν γίνει το άτυπο συμβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Merci, Ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουν ορισμένε λεπτομέρειε, όμω είπατε και σήμερα το πρωί ότι ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε ακριβώ. Δεν είναι εδώ ο κύριο Κολμέρ, κυρία Δελιάδα, ούτε, ούτε ο κύριο Ομαζή. Ο κύριο Βάλια έχει το λόγο, παρακαλώ. Α, για τους πράσινους. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Σολέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, εξ ονόματος ε, της Ελγα Τρούπολ, της Γεώδους Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές για τα όσα έχουν κάνει και για τη βούλησή τους ε, για εξέβρεση συμβαστικών λύσεων. Είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την επίτευξη μιας ισχυρής και ευρεία συμφωνίας για τους ίδιους πόρους μεταξύ των φιλευρωπαϊκών δυνάμεων και νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία. Ως πολιτική ομάδα είχαμε θέσει ορισμένες προτεραιότητες για τις διαπραγματεύσεις Πρώτον, θέλουμε να μειώσουμε ε, το μερίδιο των εθνικών συνεισφορών στο ευρύτερο σύστημα ιδιών πόρων. Και γενικά συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες. Δεύτερον, όχι πια εκπτώσεις. Και αυτό το έχουμε καταφέρει. Και τρίτον, να καταρτήσουμε έναν κατάλογο νέων ιδιών πόρων που να είναι φιλόδοξος. Και είμαστε σε θέση να πετύχουμε και αυτό το στόχο. Συνολικά λοιπόν μας ικανοποιεί αυτή η έκθεση. Θα συμμετάσχουμε και θα υποστηρίξουμε του, τις περισσότερες συμβαστικές λύσεις και από εδώ και πέρα Ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστούν οι προτάσεις μας και θα ενταχθούν στο νέο σύστημα ιδίων πόρων ε, στο ευερχόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Βάλλη. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τους δύο εισηγητές για την μεγάλη προσπάθεια που έκαναν, για τον τρόπο που δούλεψαν και τους υπόλοιπους και ηγητές να ευχαριστήσω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Λοιπόν, η δική μας θέση ως ομάδα είναι υπέρ του να αποφύγουμε τις αυξήσεις των συνεισφορών, των καθαρών εθνικών συνεισφορών, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στους προϋπολογισμούς. Ήδη υφίστανται πίεση οι προϋπολογισμοί. Ε, κάνουμε κάποια έξοδα για να τονώσουμε τη ζήτηση, που είναι σημαντικό για να υποστηρίξουμε την απασχόληση και την οικονομική ανάκαμψη στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, θα πρέπει να αποφύγουμε να βάζουμε μέτρα ε, φορολογικά, τα οποία πιέζουν και συμπιέζουν και, και ακυρώνουν ας πούμε, τη ζήτηση και πλήττουν τομεί. οι οποίοι όμως είναι πολύ ενδιαφέροντες. Ε, και οι οποίοι τελικά δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Επίσης, να βρούμε μια λύση για, τη, ε, για, τους, για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Αυτά τα εξετάσουμε και στην ΕΚΟΝ, στην Οικονομική Επιτροπή. Ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ενιαία αφαιρολογική βάση ένα μέρο από τα έσοδα αυτά πρέπει να πηγαίνει στον κοινοτικό προπολογισμό. Πρέπει να βρούμε λοιπόν το σωστό συμβιβασμό για το πώ θα εφαρμόσουμε την ενιαία αφρολογική βάση και πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ποσά αυτά, ούτω ώστε να μην υπάρχουν υπερβολικέ συνεισφορέ από, από του εθνικού προπολογισμού. Σε περίπτωση που προσθέτουμε διάφορες, διάφορους φόρους, συναθρίζουμε διάφορους φόρους. Η θέση μας λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε επικοδομητικό πνεύμα, να συνεργαστούμε στους συμβιβασμούς και τελικά θα πάρουμε μια απόφαση με βάση τις, τις δικές μας πολιτικές θέσεις εννοείται. Merci. En absence... Ευχαριστούμε. Δεν είναι εδώ ο κύριος Κολμέν, που είναι σκιώδης συζητητής. Ο κύριος Κιουσμούγκ έχει το λόγο, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές για το σχέδιο έκθεσης. με την οποία έχουμε καταλήξει ορισμένε συμβαστικέ προτάσει, θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία. Ε, η πρόταση κατάργηση των εκτόσεων σε σχέση και με το Brexit σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε. Ελπίζουμε η λύση αυτή να περάσει και στο Συμβούλιο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι θα ήταν καλό να έχουμε μια ευέλικτη προσέγγιση σε ό,τι αφορά ε, τις νέες κατηγορίες ιδίων πόρων. Και εδώ έφεσα την προσοχή σας στο γεγονός ότι οποιαδήποτε πιθανή πρόταση που ε, έχει να κάνει με περιβαλλοντικά τέλη απαιτεί κάποιο είδους ε, αντιστάθμισμα από πλευράς δαπανών. Η προσέγγιση που παρουσίασε ο κύριος Λεβαντόφσκι προηγουμένως λοιπόν θα πρέπει να λεφθεί σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν όλες τις πολιτικές ομάδες και τους εισηγητές και τους σκιώδεις. Ποιος άλλος θα να πάρει το λόγο. Για τα όσα έχουμε ακούσει. Από ό,τι βλέπω κανείς. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπα πριν. Αν υπάρχει κοινό εταιρικό φόρο, θα πρέπει, θεωρώ, να λάβουμε υπόψη και τις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργήσει αυτό όταν έχουμε λίγες εταιρείε και, πολλού και πολλούς φόρους Ο κύριος Δεμπχέμ, ευχαριστώ. Για το τελευταίο αυτό σημείο, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν αποτελεί αρμοδιότητα της δική μα επιτροπή, αλλά το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι άλλοι συνάδελφοι, ο κύριος Λαμασούρ, ε, θα υποβάλει έκθεση για τον άξονα αυτό που προανέφερα και ε, σίγουρα έχει λάβει υπόψη και τα στοιχεία που μόλις θίξατε κι εσείς. Συνολικά χαίρομαι ιδιαίτερως ε, για την στήριξη που δείξατε στο αποτέλεσμα των εργασιών μας. Είναι σαφές ότι οι επιλογές που αναφέρονται στην έκθεσή μας είναι ξεκάθαρες, ούτε ε, έκπτωση, ούτε έκπτωση στην έκπτωση, φεύγουν, εξαφανίζονται αυτοί οι μηχανισμοί για το ερώτημα του συναδέλφου, ιδίω ότι φορά τον περιβαλλοντικό κλάδο που θα φυγεί περισσότερο από ό,τι άλλοι, ε, αναφέρεται ρητός ότι μία έκπτωση ε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μόνο ένας μηχανισμός που θα μπορούσε μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων αυτό είναι μια δυνατότητα που αναφέρεται ρητός ε, στην έκθεση. Ε, βέβαια χωρίς ε, υπερβολικό άχθος ε, προς τον προπολογισμό συνολικά. Και εσείς, Πρόεδρε, το έχετε τονίσει ιδιαίτερως και δικό μας μέλημα και μάλλον το δικό μας καθήκον ήταν διπλό. Και με βάση τα όσα είπε και ο κύριος Βάλη, είναι μικρά τα περιθώρια των προπολογισμών σε εθνικό πλαίσιο, οπότε είναι ένα δύσκολο εγχείρημα όλο αυτό και εμείς είμαστε αρκετά ε, επιφυλακτικοί. Προτιμούμε να στραφούμε προς τους ε, ιδίους πόρους γιατί δεν πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό φόρο και επιμένω προς αυτό. Δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό φόρο αυτό καθ' αυτό. είναι ένα τμήμα των φόρων που εισπράττονται σε εθνικό επίπεδο και θα διοχετευθούν προς τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Η αρχή λοιπόν της δημοσιονομική κυριαρχίας των κρατών μελών ε, διασφαλίζεται πλήρως. Από την άλλη, οι δικέ μας προτάσεις ε, επιτρέπουν και την εξέβριση ισορροπίας μεταξύ ιδίων πόρων που θα συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό ε, με τα στοιχεία που έχουν τους φόρους που έχουν εισπραχθεί για να προχωρήσουν μετά και με τους ίδιους πόρου που δεν θα ανέρχονται στο ίδιο ποσοστό. Λαμβάνω λοιπόν υπόψη ότι ακόμα παραμένουν κάποια λεπτά σημεία. Νομίζω όμως ότι θα καταλήξουμε σε μία φιλόδοξη αλλά και λογική πρόταση και συμφωνία. Κάτι που εκκρεμεί ακόμα και το ανέφερε ο κ. Σολέ η λογική της έκθεσης Μόντι. Ε, θέλω να το επιβεβαιώσετε κι εσείς, ότι οι νέοι ήδη οι πόροι δεν αποτελούν επιπρόσθετο πόρο ε, για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, αλλά επιτρέπουν ε, τη μείωση των εθνικών συνεισφορών στη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Κύριε Ντουπχέ. Υπάρχουν δύο αρχές, τις οποίες έχουμε προασπίσει ε, με όλες μας τις δυνάμεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέραν της πενταετούς ε, διάρκειας του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Μία είναι ακόμα ιερή, η δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών μελών. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει αυτή την αρμοδιότητα και την κύρωση των αποφάσεων για τους ίδιους πόρους. Υπάρχει μάλιστα και απαιτεί τομοφωνία στο Συμβούλιο με περιορισμένε δυνατότητε από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερον, η έκθεσή μα θέλουμε να συνάδει και με την έκθεση Olbricht Τομά. Και αν θέλουν περίπου τον ίδιο προπολογισμό πάνω κάτω, χωρί τον Ηνωμένο Βασίλειο, κάπω πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό. Είτε μέσω του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματο, είτε με ιδίου πόρου. Δεν έχουμε άλλε επιλογέ. Βάσει και τη ε, δεύτερη ε, έκθεση, που επίσης ενθαρρύνει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να, έχει, ε, να προβλέψει επαρκείς πόρους για τις δαπάνες. Πρόθεση λοιπόν είναι κάπως να καλυφθεί το κενό μετά τον Brexit. Λοιπόν, αν σας καταλαβαίνω καλά, οι νέοι ήδη πόροι δεν θα αυξήσουν το φορολογικό βάρος εκτός από το τμήμα που θα αντισταθμίσει τη μείωση της καθαρής συνεισφοράς που μέχρι τώρα συνεισφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο στον ενωσιακό προπολογισμό. Ο κύριος Δεπρέ. Ναι, λέει ο κύριος Δεπρέ, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που μόλις είπε ο συνάδελφος Γιάννους Λεβαντόφσκι όπως ακριβώς το λέμε σαφέστατα στην έκθεσή μας. Ο στόχος μας δεν είναι λοιπόν να αυξηθεί το φορολογικό βάρος, γνωρίζοντας ότι εάν τα κράτη-μέλη με τη δική μας συμφωνία, μετά από πρόταση της Κομισιόν κτλ, εάν αποφασίσουν να ανταποκριθούν σε μια σειρά από νέε προκλήσεις, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, το θέμα είναι ποιο τμήμα των δαπανών των κρατών μελών που θα μπορέσουν να μειωθούν λόγω των επενδύσεων που θα κάνουμε σε αυτές τις νέες πολιτικές. Ο στόχος λοιπόν είναι να καταλήξουμε σε αυτό που λέτε. Αλλά ίσως κάποια στιγμή, κατά τη μεταβατική περίοδο, που δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, κανείς δεν μπορεί να την καθορίσει μέχρι τώρα, θα πρέπει να αντισταθμίσουμε και το κενό του Brexit. Και να δούμε να, θα μπορέσουν να μειωθούν διαρθρωτικά οι δαπάνες όταν θα γίνει ε, πραγματικότητα μεταφορά και πόρων και αρμοδιοτήτων. Δηλαδή θα ζητήσουμε λίγο περισσότερο φόρο, αλλά όχι περισσότερο από του φορολογούμενου. Ναι, λέει ο κύριο Ντεπρέ. Εάν είμαι αισιόδοξο, θα μπορούσα να το πω έτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είχα ζητήσει το λόγο, γιατί εκφράστηκε η ομάδα μου αλλά άκουσα τη συζήτηση και μπορεί να υπάρχουν κάποιες συγχύσεις. Νομίζω όμως ότι τώρα τα εξήγησε καλά ο κ. Ντεπρέ. Το επίπεδο δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίπεδο αυτό το καθορίζει το πουδουπού, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ανεξάρτητα από τη σύνθεση των ιδίων πόρων, έτσι. Το πολιετές πλαίσιο, ανεξάρτητα από το αν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, αυτό είναι άλλη απόφαση. Η ήδη οι πόροι θα προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του πουδουπού. Εμείς για τους ίδιους πόρους προτείνουμε να έχουμε άλλους πόρους, πιο σημαντικούς, που να μην είναι εθνικές συνεισφορές και να δούμε τι ισορροπία θα προκύψει ανάμεσα στις εθνικές συνεισφορές και αυτούς τους νέους ιδίους πόρους υπέρ του προπολογισμού της Ένωσης. Από την έκθεση όμως για τους ιδίου πόρους δεν ξέρουμε αν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Έτσι, από αυτό δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, δεν το ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή, να το πούμε με άλλα λόγια, λέει ο Πρόεδρος. Θα έχουμε ίδιους πόρους, νέους ή όχι. Ο, ανεξάρτητα από αυτό, οι δαπάνες δεν αλλάζουν, είναι ίδιες. Και το θέμα είναι πώς θα αντισταθμίσουμε τις απώλειες λόγω του γεγονότος θα, θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι καθαρός εισφορέας. Έτσι. Θα δούμε τι θα συμφωνηθεί για όλες τις δαπάνες, τις συνολικέ δαπάνες και με βάση αυτό θα πρέπει να βρούμε πόρους. Τώρα, και αν ε, υπάρξουν νέοι ήδη πόροι, θα αφαιρεθούν αυτοί από τις εθνικές συνεισφορές. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να συνεισφέρουν τα ίδια και περισσοτερα κρατημέλη. Αντίθετα, αν υπάρχουν νέοι είδη πόροι, θα συνεισφέρουν λιγότερο τα κρατημέλη. Πολύ ωραία. Μπορούμε να σταματήσουμε εδώ τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους τότε νομίζω ότι θα υπάρχει μια πλατιά συμφωνία με βάση τους συμβιβασμούς και θα ψηφίσουμε, φαντάζομαι, με ένα τέτοιο τρόπο που οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε με την έκθεση. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην εξέταση του Πουδουπού μετά το 2020. Θα το επόμενο λοιπόν πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ποιος θέλει να ξεκινήσει να κάνει τον με η κυρία Τομά, ο κύριος Όλμπριχτ. Η κυρία Τομά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλες τις ομάδες που συνεισέφεραν σε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε μπροστά μας, τους συναδέλφους καταρχάς, τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους συναδέλφους, γιατί όλοι συνεισέφεραν με 683 τοπολογίες και 75 συμβιβασμού. Ευχαριστώ όλες τις ε, ομάδε τη Επιτροπή προπολογισμού και τι πολιτικέ ομάδε και του ε, εισηγητέ και σκιώδεις εισηγητέ που έκαναν θαυμάσια δουλειά σε χρόνο ρεκόρ. Δεν θέλαμε να πούμε στον Κίνες, δεν δουλέψαμε γι' αυτό για να πούμε στον Κίνες, αλλά για να είμαστε έτοιμοι πριν από την συνεδρίαση του Συμβουλίου την Παρασκευή. Ήταν ένα πολιτικό στόχο πολύ σημαντικό ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να είναι το πρώτο όργανο που θα δώσει τη θέση του και θα θέσει τον τόνο για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επομένως, για το οικονομικό μέλλον της Ένωσης. Κάνω το σταυρό μου. Δεν ξέρω ακόμα, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε, γιατί θα ψηφίσουμε κανονικά αύριο αυτή την έκθεση, που είναι πάρα πολύ σημαντική και που θα δώσει μια εντολή διαπραγμάτευσης στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, με βάση αυτή την έκθεση, μισό λεπτό, με λιγάκι, ψάχνω τα λόγια μου, θα γίνει η διαπραγμάτευση. Και θα συζητήσει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Έτσι θα πρέπει να δείτε αυτή την έκθεση πάντως. Κάτι άλλο τώρα. Ούτω ώστε να είναι χρήσιμη αυτή η εντολή διαπραγμάτευσης. Δεν θέλω να μπω σε όλου τι λεπτομέρειε των συμβασμών, αλλά για να είναι χρήσιμη αυτή η εντολή θα πρέπει και το Συμβούλιο να μα δώσει, να μα κάνει ένα μήνυμα, να μα στείλει ένα μήνυμα. Αύριο θα ξέρουμε ποια θα είναι η τελική θέση τη επιτροπή Προπολογισμών. Μετά από αυτή τη θέση θα πρέπει να επιμείνουμε αρκετά, ούτω ώστε το Κοινοβούλιο να συζητήσει με το Συμβούλιο. Χθε στην ε, Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση η παρουσία της Βουλγαρικής Προεδρίας ε, στείλαμε τον μπαλάκι στο Συμβούλιο και του είπαμε ότι περιμένουμε τον εκπρόσωπο της ε, Προεδρίας, της Βουλγαρικής Προεδρίας που είχαν προβλέψει δύο συνεδριάσεις το μήνα μεταξύ του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Αυτό μας είπαν και τους είπαμε εμείς, ε, κοιτάξτε, εμείς προς το παρόν δεν βλέπουμε να έχετε προβλέψει τίποτα μαζί μας. Το επαναλαμβάνω βεβαίως, ξέρω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής εδώ το ξέρουν, ότι τελικά θα πρέπει να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας ή να μην τη δώσουμε. Επομένως και τα δύο όργανα, και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχουν κάθε συμφέρον να αρχίσουν κοινέ συζητήσεις των συντομότερο δυνατόν. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Κλείνοντας θέλω να πω ότι βρήκαμε ισορροπίες βάζοντας 75 συμβασμούς μέσα στην έκθεση αυτή. Βάλαμε πολλούς συμβιβασμούς. Μοιάζει λιγάκι με τη συζήτηση που έγινε για τους ίδιους πόρους. Ένα συμβιβασμό δεν σημαίνει ότι όλοι μας είμαστε 100% ικανοποιημένοι. Προφανώς υπάρχουν σημεία τα οποία κάποιοι επιθυμούν περισσότερο, κάποιοι άλλοι λιγότερο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Αλλά είναι πολλοί οι συμβιβασμοί. Και αυτοί οι συμβιβασμοί προφανώς έχουν σαν στόχο να δείξουν ότι είναι ενωμένο το Κοινοβούλιο σε αυτή τη συζήτηση με το Συμβούλιο. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι, ότι υπάρχει ενότητα εδώ, τουλάχιστον πιο πολύ από το Συμβούλιο. Είμαστε λοιπόν σε ισχυρή θέση και αυτό είναι καλό μην πω ότι είμαστε και πιο ενωμένοι από την Κομισιόν. Ενώ έχει θεσμική υποχρέωση να δείξει ενιαίο πνεύμα. Δείτε τι είπε ο κύριος Έτιγκερ και ο πρόεδρος Γιούνκερ την περασμένη εβδομάδα. Δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη στάση σας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε αυτή την ενωμένη στάση. Ήθελα, ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά το ξεχνάω τώρα. Δεν πειράζει. δεν τελείωσαν οι ευχαριστίες, γιατί είμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Παρότι έχουμε, μοιάζει να τελειώσαμε κάτι, στην πραγματικότητα τι τελειώσαμε. Τελειώσαμε την, ολοκληρώναμε εδώ δηλαδή την εντολή διαπραγμάτευση. Τώρα αρχίζουν τα υπόλοιπα. Α, θυμήθηκα τι ήθελα να πω. Μετά από αυτά που είπε ο κύριο Ντεπρέ και ο κύριο Λεβαντόφσκι. Θα επιβεβαιώσουμε ότι η έκθεση για τους ίδιους πόρους και το πουδουπού, το πολυδές δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, και θα το επιβεβαιώσει ο κύριος Έλμπριχ, είναι πράγματα που πάνε χέρι-χέρι. Έτσι, είναι δύο εκθέσεις που πάνε χέρι-χέρι. Και να χαιρετήσω πολύ φιλικά και θερμά το συνεισηγητή μου, τον κύριο Όλμπριχτ, με τον οποίο ήταν μια απόλαυση η συνεργασία και θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία ε, στα πλαίσια τη διαπραγμάτευση μέσα στο 18. Ε, χαιρόμαστε που σα τόσο ευτυχή, Ιζαμπέλ, που συνεργαστήκατε με τον κύριο Όλμπριξ, στον οποίο δίνω και το λόγο. Μίλησε προηγουμένω για το ρεκόρ Guinness. Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποια, έκανε έτσι υπενιγμούς προς την αποστολή σας ε, στην Ιρλανδία. Γι' αυτό νομίζω ότι πάντα είναι πολύ αποτελεσματικέ οι αποστολέ τη ε, Επιτροπή μα και αυτή τη φορά ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Δουλέψαμε ακόμα και η ισότητα των φύλων ε, υπήρχε και είχε καλυφθεί με καλή ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και εγώ αρχικά να σταθώ στο έργο της ε, συνεισηγήτριας που είναι πραγματικά πολύ αποτελεσματική, παρότι δεν ήταν εύκολο καθήκον λοιπόν. Έχουμε εργαστεί επί των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να προσθέσω όμως ορισμένες παρατηρήσεις. Σκοπός μας ήταν ε, η εξέβρεση συμβαστικών λύσεων σε περιπτώσεις όπου ήδη έχουμε ζητήσει την γνωμοδότηση εξειδικευμένων επιτροπών που έχουν θεσπιστεί όχι μόνο για την έκθεση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και για τη συζήτηση ε, για, συγκεκριμένα για τους κανονισμούς. Δεν μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη όλες τις λεπτομέρειες ε, των ε, εκθέσεων των νομοδοτήσεων των εξειδικευμένων επιτροπών, γιατί αυτό παρεμβαίνει και στις μελλοντικέ τομεακές πολιτικές. Νομίζω θα τα λάβουμε αυτά υπόψη στο μέλλον και είναι χρήσιμο για να κατανοήσουμε αφενός ε, την γενική θέση ε, αυτής της Επιτροπής για το Πίδελταπή και για να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Στη δική μας έκθεση έχουμε ορισμένα γενικά στοιχεία και τη δομή του επερχόμενου Πίδελταπή, αλλά για κάποια συμπεράσματα σχετικά με επιμέρους πολιτικές. Έχουμε συμπεριλάβει τα κύρια στοιχεία. Και ε, συναντηθήκαμε και με τους ε, εισηγητές των νομοδοτήσεων, αλλά και με τους σκιώδεις. Προσπαθήσαμε και βρήκαμε, θεωρώ, τον ε, τρόπο να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που ικανοποιούν τουλάχιστον και τους ασκιώδεις ηγητές. Υπάρχουν και δύσκολα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι και πάλι καταλήξαμε σε συμβαστικέ λύσεις. Υπάρχουν βέβαια και στοιχεία που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε συμβαστικέ λύσεις, αλλά αυτό πάντα συμβαίνει όταν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές απόψεων. Εν γέννη, συμφωνούμε επί των προτεραιοτήτων, επί του επίπεδου ε, του προπολογισμού έχουμε συμφωνήσει και για τη δομή, ακόμα και αν δεν συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες με την αλλαγή της δομής, γιατί υπάρχει αυτή η επιλογή, είτε θα αλλάξουμε δομή είτε όχι. Εμείς προτείνουμε να αλλάξουμε, αλλά και όχι τόσο επαναστατικά τη δομή του προπολογισμού δείξαμε και ορισμένα στοιχεία για τη διασύνδεση μεταξύ των μέρους πολιτικών και προσπαθήσαμε να βρούμε ε, συμβιβασμού για συγκεκριμένα ζητήματα που είναι εξαιρετικά δύσκολα, όπως η αιρεσιμότητα. Όπως έχει προταθεί από πολλούς συναδέλφους. Κλείνοντας, νομίζω ότι αυτή η εκδοχή που προτείνεται αυτή τη στιγμή είναι αυτή στην οποία καταλήξαμε και καταφέραμε να πετύχουμε μαζί με τους αισθιώδεις εισηγητές. Και ευχαριστώ όλη την ομάδα που εργάζεται μαζί μας γιατί είναι πραγματικοί επαγγελματίες και πολύ άξιοι. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που δυσκολεύουν ορισμένου, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε, και είναι σημαντικό να έχουμε την κοινή θέση του Κοινοβουλίου. Και τέλο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται σε δύο ημέρε. Εμεί ψηφίζουμε αύριο. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε στο Συμβούλιο. Εντάξει, βέβαια είναι μόνο η Επιτροπή μα δεν είναι ολόκληρο το Κοινοβούλιο, αλλά και πάλι. Είναι σημαντική και αυτή η στάση. Να δείξουμε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι έχουμε ξεκάθαρη και ισχυρή θέση. Και είναι σημαντικό να αποστείλουμε αυτό το μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να είναι σαφές λοιπόν ότι τελικά η θέση μας θα είναι αυτή που θα καθορίσει το αποτέλεσμα, θα πούμε ναι ή όχι. Πλέον έχουμε και δικαίωμα να πούμε όχι λοιπόν. Γι' αυτό θέλουμε να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις. Γιατί πάντα υπάρχει πιθανότητα να απορρίψουμε την μελλοντική πρόταση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βιαστούμε και να προετοιμαστούμε εγκαίρως και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε λοιπόν για κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο για την ε, εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Πράγματι, πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε και να εμπνεύσουμε και τους ε, αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων που ε, θα συζητήσουν την Παρασκευή και αυτό το θέμα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και είπατε πολύ σωστά ότι για μας δεν έχουμε αφενός τους νέους ιδίους πόρους και αφετέρου το ΠΔΠ. Πρόκειται για ένα ενιαίο και αδιέρετο σύνολο. Και μετά για το κατά πόσο έχουμε δικαίωμα να πούμε ναι ή όχι, αυτό σημαίνει ακριβώ ότι θα πρέπει ευθύ εξ αρχή να συμμετάσχουμε ε, στις διαπραγματεύσει μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ακούσαμε και τους ασκιώδεις συζητητές. Έχουμε ένα σχέδιο συμβιβασμού που θεωρούμε ότι ε, θα τύχει ευρεία στήριξη στην Επιτροπή μας οι ομάδες του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών Δημοκρατών έχουν ε, εκπροσωπηθεί λοιπόν. Ο κύριος Κολμέλ, ο κύριος Κισμούκ θέλει να μας ε, παρουσιάσει τη θέση των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τους συζητητές για την έκθεση. Είμαι μέλος της ε, Επιτροπής Γεωργικών Υποθέσεων. Θα ήθελα λοιπόν ε, να επισημάνω δύο θέματα εδώ που έχουν να κάνουν με τη Γεωργία. Θα ήταν καλό να συμπεριλάβουμε και μια διάταξη που να αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξει ε, ισοστάθμιση των πληρωμών για όλα τα κρατημέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει ίσο παιδί ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Έχουμε υποβάλει και εμεί μια τέτοια τροπολογία, ελπίζω να ληφθεί υπόψη. Άλλο εξίσου σημαντικό θέμα. Προτινόμενες αλλαγές σε ορισμένα τμήματα του προπολογισμού είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τις ε, δαπάνες ε, για τη γεωργία Ω ένα ξεχωριστό τμήμα του προπολογισμού. Βέβαια αυτό έχει επιπτώσεις και σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Εάν καταργηθούν αυτά τα τμήματα, αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τι ε, μελλοντικέ ε, δαπάνε. Αυτέ ήταν οι δύο επισημάνσει που θέλω να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ντεπέ. Ευχαριστώ πρόεδρε όπως και όλοι οι συνάδελφοι εκτιμώ ιδιαίτερα την ποιότητα της εργασίας των δύο συνεισηγητών μας και ε, επίσης την προσπάθεια που έκαναν για να επιτύχουν ε, συμβασμούς. Υπάρχουν τρία βασικά θέματα με τα οποία συμφωνούμε πλήρως με την πρόταση που μας έχει υποβληθεί. Το πρώτο Πρέπει να έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για να καλύψουμε τις πολιτικές που εμείς οι ίδιοι αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε, να εκτελέσουμε. Δηλαδή, εάν για να καλύψουμε τις πολιτικές χρειάζεται το 1,3 του ΑΕΕ, τότε πρέπει να ζητήσουμε το 1,3 του ΑΕΕ. Επίσης, οι προτεραιότητες που προτείνονται σε αυτό το κείμενο είναι σαφείς και οι δυνατότητες ε, ευελιξίας μας επιτρέπουν να υπάρξουν οι αναγκαίες ε, αυξήσεις αν χρειαστεί και στα ποσά και στο ποδίο εφαρμογή. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις πολιτικές που θεωρούμε ουσιώδεις. Αλλά όπως επιθυμούν οι περισσότερες ομάδες θα πρέπει να διατηρηθούν τα βασικά κεκτομένα στα βασικά συγγνώμη, και εκτιμένα τη κοινή γεωρική πολιτική και τη πολιτική σύνοχή. Βεβαίω, για παράδειγμα, ο ε, ορίζον 2020, σύν μικρομεσαίε επιχειρήσει, όλα αυτά. Και με χαρά σημειώσαμε ότι οι συνεισηγητέ θέλουν να ληφθούν τα μέτρα που προκύπτουν από την COP21. Επίσης, μας ικανοποιεί η επιθυμία που εκφράζουν να μην υπάρξει ε, ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός εξωτερικών μέσων χρηματοδότησης του προπολογισμού που διαφεύγουν από κάθε κοινοβουλευτικό έλεγχο υπόλων. Αυτό λοιπόν έχετε την συμφωνία μας. Τώρα υπάρχουν κάποιες δυσχέρειες. Θα αναφέρω μία, γιατί την ανέφερε και ο κύριος Όλμπριχτ. Δεν θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να μελετήσουμε τη δομή. Οποιαδήποτε δομή και αν προταθεί δεν θα μας βρει σύμφωνος. Δεν νομίζουμε ότι είναι το βασικό στοιχείο της συζήτησης. Τώρα, κάποια άλλα σημεία που μας ενοχλούν και τα οποία προκαλούν μεγάλες συζητήσεις στο εσωτερικό της ομάδας μας. Πρώτον, διάρκεια του ΠΔΠ. Συνολικά η ομάδα μας είναι υπέρ πενταετούς πει και όχι επταετούς όπως προτείνεται. Σας το λέω γιατί αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Ανεξάρτητα από την προσωπική μου άποψη πρέπει να σας ε, ενημερώσω για την ε, πλειοψηφική άποψη της ομάδας μου. Δεύτερον, ε, πιο λεπτό και αυτό προκαλεί συζητήσεις και επί του οποίου η ομάδα μου δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Τώρα τελευταία διατυπώθηκε εξή άποψη. Μα καλά. Θέλετε να υπάρξει συμφωνία για τα 7 επόμενα έτη επί ενός πι με βάση αυτά τα δύο στοιχεία. Εάν θέλετε να συμφωνηθεί σύντομα το πι πι, θα το κάνετε όσο θα είναι ακόμη θα συμμετέχουν οι Βρετανοί. Για μια περίοδο κατά την οποία δεν θα συμμετέχουν. Σας εξηγώ τι λένε κάποιοι και τι συζητιέται στην ομάδα μου για να καταλάβετε. Για να μην πείτε ότι μετά δεν ε, σας έχουμε ενημερώσει για το τι μπορεί να προκύψει. Λέει αυτή η άποψη. Μα είναι σκόπιμο και σε κοινοβουλευτικό και σε επίπεδο συμβουλίου να συναποφασίσουν όχι μόνο στις κατευθυντήριες γραμμές αλλά και να συναποφασίσουν το ίδιο το ΠΔΠ που δεν θα του αφορά πλέον. Πρώτο στοιχείο αυτό. Δεύτερο, που συνδέεται το επόμενο κοινοβούλιο που θα εκλεγεί το 19. Είναι δυνατόν να έχει δεμένα τα χέρια από προηλημένες αποφάσεις, να μην έχει καμία δυνατότητα να τροποποιήσει την κατάσταση. Η ομάδα μας κάνει μια μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αλλά θέλω να ενημερωθούν οι άλλοι συνάδελφοι. Άρα και για τη διάρκεια και για τη στιγμή έγκριση του ΠΔΕΛΤΑΠΗ, αυτά τα δύο στοιχεία λοιπόν προκαλούν πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό της ομάδας μου. Για το περιεχόμενο, με την εξαίρεση κάποιων, λεπτομεριών, ιδιαίτερα τη δομή, υπάρχει αρκετά ευρεία συνένεση, αλλά αυτά τα δύο στοιχεία που ναι, είναι συγκυριακά αλλά δεν είναι μικρή σημασία, αυτά τα δύο σημεία ε, προκαλούν μεγάλη ζήτηση στο εσωτερικό της ομάδας Άλντε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα. Ε, τώρα δεν βλέπω εκπρόσωπο της Γκουα, οπότε ο κύριος Σολέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αύριο πρωί Έχουμε την άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου από αυτού. Άρα έχουμε την ευκαιρία ως Επιτροπή να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη. Το οποίο θα πρέπει να είναι. Όχι και άλλες περικοπές. Όπως ε, επανειλημμένα έχετε πράξει. Έχουμε πολλές προκλήσεις ενώπιών μας. πολλές ανάγκες να καλύψουμε και θα προκύψουν και απρόβλεπτα. Άρα το ΠΔΠ πρέπει να είναι φιλόδοξο να μπορεί να αποκριθεί σε όλες αυτές τις αναμενόμενες αλλά και απρόβλεπτες προκλήσεις. Για την ομάδα μας υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να πούμε στα κράτη-μέλη από πλευράς προτεραιοτήτων. Η Ένωση πρέπει να τιμήσει τις διεθνείς θεσμεύσεις της, ιδιαίτερα για τους βιώσιμους στόχους και την κλιματική αλλαγή. Για μας πρέπει να υπάρξει λοιπόν σαφής αναφορά της συμφωνίας των Παρισίων και των στόχων επί των οποίων έχουμε δεσμευθεί. Εντάξει, βέβαια, οι συμβαστικέ διατυπώσει ε, ποτέ δεν μπορούν να ικανοποιούν τι αρχικέ ε, επιδιώξει όλων. Αλλά το στόχος του 30% των δαπανών να συνδέονται με την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής δεν είναι αυτός που θα θέλαμε, δεν ήταν η αρχική μας θέση, αλλά είναι συμβαστική πρόταση, μπορούμε να τη στηρίξουμε. Είναι ένα καλό βήμα προς τα μπρος. Βέβαια υπήρξαν πολλές τροπολογίες, άρα και πολλές συμβαστικές. Κάποιες δικές μας τροπολογίες ε, ελήφθησαν υπόψη, άλλες όχι. Άρα δεν συμφωνούμε επί όλων. Δεν συμφωνούμε για τις δαπάνες για την άμυνα, ούτε για τον πυρηνικό τομέα, ούτε για την αποθήκευση του άνθρακα. Λυπούμεθα που δεν υπάρχει πρόταση για να γίνουν έστω και κάποιες μικροαλλαγές σε σημαντικές πολιτικές όπως η γεωργική, η πολιτική συνοχής όπου είχαμε υποβάλει κάποιες προτάσεις, οι οποίες ε, δεν ελήφθησαν υπόψη στις συμβιβαστικέ. Και υπάρχουν και άλλες συμβαστικές προτάσεις, των οποίων το περιεχόμενο ακόμη το συζητάμε ως ομάδα. Για παράδειγμα για την αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου. και για τη νέα δομή του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Αλλά συνολικά και επειδή υπάρχει και μεγάλη πίεση, τρομερή πίεση χρόνου, δηλαδή εργαστήκαμε υπό τρομερή πίεση χρόνου επ' αυτών των συμβαστικών, νομίζω ότι η τελική έκθεση θα είναι καλή και θα στείλει σαφή και ηχηρά μηνύματα προς τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη επιμονή και συνέπεια στην υπεράσπιση των θέσεών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάλλη δεν είναι εδώ, άρα το EFTD δεν θα εκφραστεί και ούτε και το ENF. Λοιπόν, τώρα ποιοι άλλοι συνάδελφοι πέραν των σκιωδών θέλουν το λόγο. Ο κύριος Ρίμπιχ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Από την αρχή της συζήτησης το βασικό πρέπει να είναι το χρονοδιάγραμμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Κοινοβούλιο μέσω της εργασίας των βουλευτών και των υπηρεσιών μας είναι καλά προετοιμασμένο και έχει εντοπίσει τα βασικά προβλήματα και κατέληξε σε καλές συμβαστικές προτάσεις. Εάν δεν εγκριθεί διαδικασία fast track, το Συμβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται με το συνήθι ρυθμό του δεν βιάζεται και θα περιμένει να προκύψουν νέοι βουλευτές, ε, νέοι πρόεδροι, νέοι επίτροποι και το Συμβούλιο με την ησυχία του κατά την Κροατική ενδεχομένως Προεδρία θα καθορίσει ένα νέο πρόγραμμα. Οπότε εμείς ε, θα πρέπει να πιέσουμε για να γίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Και θα θέλαμε στα συμπεράσματα και στα πρακτικά του Συμβουλίου Κορυφής να εγκριθεί αυτή η ταχεία διαδικασία, fast track. Γιατί έτσι θα είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί. Ιδιαίτερα για το ένα το πρόγραμμα έρευνας είναι απολύτως αναγκαίο. Γιατί μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από τη μία και επειδή ακούγεται ότι η μεταβατική περίοδος ε, ε, δεν θα έχει καθορισμένο τέλος, όλα αυτά δημιουργούν ε, ασάφειες. Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε το περιεχόμενο και κατόπιν εντάξει τις πιστώσεις θα τα δούμε, θα τις δούμε σε κάθε συγκεκριμένη γραμμή για να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο. Χαίρομαι που προβλέπονται τουλάχιστον 120 δις Ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο ήθελε στην ουσία διπλασιασμό για αυτό το νέο πρόγραμμα. Γιατί αν διαβάσει κανείς τις δημοσκοπήσεις ε, στο Ευρωβαρόμετρο θα δείτε ότι το πρόγραμμα για την έρευνα θεωρούν ότι είναι το καλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι σαφές λοιπόν το μήνυμα των συμπολιτών μας. Ο διπλασιασμός ή τουλάχιστον 120 ε, βάση περιπτώσει θα ήταν ένας καλός συμβασμός για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από τη συνέχιση των ε, υφισταμένων προγραμμάτων θα πρέπει να συζητήσουμε και νέα προγράμματα. Από τις δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου ξέρουμε τι αναμένει από μας ε, η κοινή γνώμη κυβερνοασφάλεια, ασφάλεια των επικοινωνιών, πρέπει να καταστεί σαφές ότι χρειάζεται φρέσκο χρήμα για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις των ε, συμπολιτών μας. Ξέρω ότι οι καθαροί συνεισφορείς δεν θέλουν να πληρώσουν κι άλλα. Οπότε δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Ο δικός μου υπολογισμός είναι ότι θα έχουμε και ένα μείον 12% λόγω του Brexit. Αλλά θα μπορούσαμε να προωθήσουμε μέσω νέων πόρων νέα προγράμματα. Για παράδειγμα στη Γεωργία. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες στις παγκόσμιες αγορές να σπάσουμε τα ολιγοπόλια ορισμένων προμηθευτών έχουμε πολύ υψηλέ δυνατότητες στη γεωργία, μέσω χρήσης ρομπότ, μέσω αυτοεκπαιδευμένων μηχανών μπορούμε πολλά να επιτύχουμε. Το ίδιο και για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τις μεταφορές, ε, για τη γεωργία. Πολλά μπορούμε να επιτύχουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέα προγράμματα. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό. Και παρακαλώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να την έχουμε στο κέντρο της προσοχής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Χωσέ Μανουέλ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τους δύο συνεισηγητές, την κυρία Τωμά και τον κύριο Ολμπριχτ, για όλα όσα έκαναν. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα για το τι πρέπει να είναι η Ευρώπη και τι θέλουμε για την Ευρώπη και να δώσουμε και ε, ένα παράδειγμα έτσι, ενότητας. Είμαστε 751 51 ευρωβουλευτές και νομίζω ότι η πλειοψη... αν δείξουμε ότι είμαστε μια μεγάλη, μια πλατιά πλειοψηφία, θα μπορούσαμε να εμπνεύσουμε τα 28 κράτη, τουλάχιστον τα 27. Να τα εμπνεύσουμε, γιατί δεν μπορώ να πω να τα υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Το θέμα του χρονοδιαγράμματος το θέμα της πενταετίας. Πολλές φορές κάναμε αυτή τη συζήτηση. Ορισμένοι λένε ότι το επόμενο κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει, γιατί αυτό έχει την νομιμότητα. Τότε να σταματήσουμε να συζητάμε, γιατί η παρούσα Κομισιόν δεν έχει τότε την αρμοδιότητα να παρουσιάσει ένα πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που θα δεσμεύσει ουσιαστικά την επόμενη Επιτροπή. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η Επιτροπή καθυστέρησε να υποβάλει την πρότασή τη. Έπρεπε να την είχε υποβάλει μέσα στο 17 κανονικά. Αλλά θέλουμε, αν θέλουμε δημοκρατική νομιμοποίηση, ποιο μα τη δίνει, η προτεραιότητα Ευρωπαϊκή Ένωση, η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, το θέμα τη εκπαίδευση και τη επαγγελματική κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτομία, η καταπολέμηση τη φτώχεια, τι θα κάνουμε, δεν θα τους υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Υπάρχουν και άλλοι μάλιστα. Ασφάλεια και άμυνα. Και ζητάμε μάλιστα μια νέα γραμμή, γιατί έτσι δίνουμε τη δυνατότητα στο νέο Κοινοβούλιο και στην επόμενη Επιτροπή να κάνουν μια προσαρμογή στις νέες προκλήσεις και στις νέες προτεραιότητες. Αυτό τι είναι ευελιξία, κυρίες και κύριοι. Εξασφαλίζουμε αυτή την ευελιξία. Και ελπίζω λοιπόν ότι το Συμβούλιο θα δείξει ευαισθησία. Θα δείξει ευαισθησία απέναντι στο ότι θα έχουμε μια νέα επιτροπή και ένα νέο κοινοβούλιο που μπορούν να προσαρμόσουν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και να προβλέψουμε και ένα χρονικό ορίζοντα, μάλιστα. Αυτά γίνονται με απλό τρόπο. Έπειτα, πέντε χρόνια για να συμπίπτει το πουδουπού με την κοινοβουλευτική θητεία. Αυτό είναι το όνειρο. Μην ξεχνάτε πόσα χρόνια χρειάζομαστε για να ετοιμάσουμε μια πρόταση. Α υποθέσουμε ότι ξεκινάμε σήμερα με ένα καινούριο φρέσκο κοινοβούλιο και, και μια φρέσκια κομισιόν. Πόσο χρόνο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταθέσει την πρότασή τη, για πέστε μα πόσο χρόνο, πόσο χρόνο θέλει το κοινοβούλιο για να συμφωνήσει, για να δώσει το πράσινο φω, πόσο χρόνο θέλουν τα κράτη-μέλη για να ετοιμάσουν τι ε, συμφωνίε εταιρική σχέση. Αυτό τι σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνο να φτάσουμε στα μέσα τη θητείας και να μην έχουμε ακόμα το πουδουπού, κύριε και κύριοι. Θα είναι πενταετέ μάλιστα, το οποίο όταν το ετοιμάσουμε το πενταετές πουδουπού, θα είναι έτοιμο για του επόμενου όχι για μα. Είναι αδύνατο να συμπέσει η δική μα έναρξη της, ε, η έναρξη της κοινοβουλευτική θητεία με την έναρξη του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αδύνατο. Επίση, θέλετε να καταργήσετε τον κανόνα νη 3 ή νη 2 γιατί τα πολιτή δημοσιονομικά πλαίσια συνδέονται. Και θέλουμε να πούμε επίσης στους πολίτες ότι το 2021 το επόμενο πουδουπού θα ξεκινήσει. Με τη φιλοδοξία που του χορηγούμε και το θέμα της ευελιξίας βοηθάει στο να δώσουμε ε, τη δυνατότητα στους επόμενους να προσαρμόσουν ανάλογα με τις επόμενες, ε, με τις προτεραιότητες που θα προκύψουν τότε. Και αυτό μας δίνει και η δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία πιστεύουμε και ελπίζουμε αύριο να συμφωνήσουμε. Είμαι για σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε, αλλά τέλος πάντων ελπίζω θα συμφωνήσουμε και στην Ολομέλεια, έτσι να δώσουμε ένα ηχηρό ναι και να συνεισφέρουμε έτσι χάρη στη δουλειά που κάνουν όλοι οι συγητές. Γιατί πρέπει να υπερψηφιστεί με πλατιά πλειοψηφία αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες απάντησε ήδη και συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε. Λέει κυρία Βάρδια Θαβάλ Ρούβιαλ. Και μία από τις ε, συζητήσεις που κάναμε εδώ στην Επιτροπή μας ήταν αυτό το αιώνιο πρόβλημα των, ε, του χρονοδιαγράμματος του Πουδουπού με την ε, κοινοβουλευτική θητεία και πώς θα συμπέσουν αυτά τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι κάθε κοινοβούλιο θέλει να έχει και φωνή και να ψηφίζει και να καθορίζει το Πουδουπού στη θητεία του. Αλλά οι ημερομηνίε είναι αυτέ που είναι. Και δυστυχώ σήμερα στο τέλος της θητεία μας θα πρέπει να αποφασίσουμε για ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί δεν το κάνουμε τώρα, θα πρέπει να το κάνει το επόμενο κοινοβούλιο. Φανταστείτε, μέχρι να συσταθεί το επόμενο κοινοβούλιο και η επόμενη επιτροπή θα είναι πολύ αργά για να μπορέσει να εγκριθεί και να μπει σε εφαρμογή όπως πρέπει. Τι να σας κάνουν, οι προθεσμίες είναι προβληματικές, αλλά αυτές είναι και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα να δουλέψουμε τώρα, ούτως ώστε να έχουμε χρόνο, παρά να δώσουμε τη σκητάλη στο επόμενο κοινοβούλιο και να καθυστερήσουμε όλα τα προγράμματα. Βεβαίως, ε, το πρόβλημα είναι, όπως είπε και ο κύριος Ντεπρέ, ότι αν το εγκρίνουμε τώρα το πουδουπού, ε, θα είναι ακόμα στο Συμβούλιο ε, οι Βρετανοί. Ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά η Βρετανική κυβέρνηση δεν θέλει να επηρεάσει και να καθορίσει τη μορφή ενός πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου στο οποίο θα συμμετάσχει. Το έχουν πει αυτό. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιεχόμενο τώρα τη έκθεσης, νομίζω ότι οι δύο εισηγητέ έκαναν μια φανταστική δουλειά, το αναγνωρίζουμε όλοι οι σκιώδει εισηγητέ και όλοι οι συνάδελφοι γενικά. Έχει πάρα πολλού συμβιβασμού η έκθεση και είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε 100% με κάθε λεξούλα, και με κάθε κόμμα και τελεία, αλλά σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να συμφωνήσουμε με του συμβιβασμού Ε, συμβασμούς που και ιδέες που εκφράζουμε οι περισσότερε πολιτικέ ομάδε καθ' όλη την ε, κοινοβουλευτική θητεία. Ειδικά οι προευρωπαϊκέ οι φιλοευρωπαϊκέ πολιτικέ ομάδε. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Λοιπόν, τι λέει αυτή η έκθεση, ότι θέλουμε να κρατήσουμε ε, τη χρηματοδότηση των παραδοσιακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν θα μπούμε στο περιεχόμενο, ε, δεν θα μιλήσουμε για τα ταμεία. Πέρα από τις τροποποίησεις που γίνονται σε αυτές τις πολιτικές, χρειάζονται κονδύλια για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και αυτό που ζητάμε είναι να κρατήσουμε αυτά τα κονδύλια. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιε πολιτικέ που μπορούμε να τι ονομάσουμε μελλοντικέ πολιτικέ που έχουν να κάνουν με την πολιτική για την νεολαία, με τι πολιτικέ ε, έρευνα και ανάπτυξη ή με την εξωτερική πολιτική, διάφορε οριζόντιε γραμμέ στον προπολογισμό επίση, που θέλουν περισσότερες, ε, περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερε επενδύσει. Γιατί είναι πολιτικέ που πάνε πολύ καλά, που λειτουργούν και όσο περισσότερα λεφτά έχουμε για αυτέ τι πολιτικέ, τόσο μεγαλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε. Τρίτον, Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι αποφασίζει το Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως το Συμβούλιο, ότι έχει νέες ε, αρμοδιότητες, νέες πολιτικές, τότε θέλουμε νέα ποσά. Δεν μπορούμε να κόβουμε, ας πούμε, κονδύλια από άλλες πολιτικές που είναι απαραίτητε. Έτσι. Και για να τετραγωνίσουμε τον ε, κύκλο, γι' αυτό φτιάξαμε και το, την έκθεση για το, τους ιδίους πόρους. Τώρα, κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, γιατί δεν υπάρχει συμβιβαστικέ τροπολογίε. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχει να κάνει τι θα κάνουμε με τα λεφτά από τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι τμήμα των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και το πρόβλημα είναι ότι παρότι έχουμε αυτά τα, αυτά έκτακτα κονδύλια, τα έκτακτα έσοδα, επειδή τα, οι παραμένουν στο ίδιο επίπεδο, τελικά αυτά τα ποσά επιστρέφουν στα κράτη-μέλη. Γιατί μειώνουμε στην πραγματικότητα τη συνεισφορά του λόγω των προστήμων. Παρότι δηλαδή έχουμε μεγαλύτερα έσοδα, αυτό δεν οδηγεί σε μεγαλύτερε δαπάνε. Δηλαδή, τα λεφτά επιστρέφουν στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω του κοινοτικού ενωσιακού προπολογισμού πηγαίνουν στι τσέπε των κρατών μελών. Έχουμε αυτέ τι τροπολογίε και προτείνουμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ούτω ώστε αυτά τα έσοδα από τα ε, πρόστιμα να μπουν σε ένα ειδικό ταμείο και να για να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποιε δαπάνε στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε κάποια προγράμματα, ας πούμε, τα οποία ξέρουμε ότι θα χρειαστούν περισσότερα λεφτά. Θα είναι ένα σύστημα του Global Margin for Commitments. Ε, του περιθωρίου που υπάρχει για τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων. Αυτά. Τίποτα άλλο. Είναι αρκετά τεχνικό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά μπαίνουν στι τσέπε των κρατών μελών. Καθώ εμεί δεν έχουμε αρμοδιότητα στα έσοδα, οποιαδήποτε επιπρόσθετα έσοδα επιτρέπουν ε, στα κρατημέλη να μειώσουν τη συνεισφορά τους. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Πρέζα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι θαυμάζω ιδιαίτερα το έργο των δύο συνεισηγητών σε συνεργασία και με τους κοιόδης συγητές και με όλους τους πολιτικούς συμβούλους και με όλη την ομάδα της Επιτροπής Προπολογισμών. Θα ήθελα παρόλα αυτά να διατηρήσουμε ένα περιθώριο ευελιξίας. Και ελπίζω να μ' ακούσει ο κύριος Φερνάντες, γιατί ο ίδιος επέμεινε σε αυτό το σημείο, καθώς και η ΕΝΤΕΡ. Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του χρόνου. Ίσως να υπάρχει μια φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι με το ΠΔΠ δεν θα παρεμποδίσουμε τις εξελίξεις μετά τις εκλογές και να αφήσουμε ένα ευρύ περιθώριο ευελιξίας. Αν πάμε πολύ παραπέρα ε, στα ζητήματα της ασφάλειας, αν τα κάτι μελη καταφέρουν πιο συλλογικά να σταθούν σε αυτά τα ζητήματα πέραν του 2019, θα μπορέσουν να μεταφέρουν κάποιες από τις ε, ε, πιστώσεις αυτές σε εθνικό επίπεδο προς το ευρωπαϊκό για να είναι πιο ε, αποτελεσματική η ευρωπαϊκή δράση στον τομέα του διαστήματος, για παράδειγμα. Γιατί αν υπάρχει ένας υπερεθνικός τομέα, αυτό είναι το διάστημα. Αλλά ο καθένα προσπαθεί να ε, προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα σε αυτό το κλάδο και την εθνική βιομηχανία. Ίσως ε, να μπορέσει να υπάρξει ε, μια πιο ξεκαθαρή τάση που θα προκύψει από τις ευρωεκλογέ και αυτό ε, θα άλλαζε και πάλι τη δυναμική των πραγμάτων. Επομένως, κύριοι συνεισηγητές, μήπως θα μπορούσαμε να αφήσουμε ένα τέτοιο παράθυρο ευελιξίας, ένα περιθώριο. Γιατί κατανοώ ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να υιοθετηθεί το στομότερο δυνατόν, για να μην έχουμε την αναστολή των εργασιών όπως το 2014, γιατί ψηφίσαμε το φθινόπωρο του 2013 το ΠΔΠ. Αλλά να διατηρήσουμε λοιπόν αυτή την ευελιξία για να πάμε πέρα από τα όσα προτείνει το ήδη φιλόδοξο ΠΔΠ, γιατί σίγουρα βέβαια πρέπει και να ε, λειτουργήσουμε προκαταβολικά γιατί γρήγορα φτάνει η πρώτη πρώτου του 2021. Πρέπει όμως να διατηρήσουμε μια ευελιξία για να μην ε, φυλακιστούμε από ένα πιδελταπή που θα έχουμε ψηφίσει πριν από τις ευρωεκλογέ και θα μας είναι στενός κορσές μέχρι το 2027 όπου σίγουρα μέχρι τότε θα ανακύψουν και απρόβλεπτες καταστάσεις και θα είμαστε υποχρεωμένοι να ιδρύσουμε καινούργια καταπιστεύματα και άλλους μηχανισμούς που θα ε, διευρύνουν και θα εντείνουν όλο αυτό το δημοσιομικό πλέγμα. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Πρέζα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο και ευχαριστούμε που είστε εδώ από το πρωί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία θα ήθελα να σχολιάσω τις παρεμβάσεις ε, και τα όσα είπαν οι συγητές. Πρώτα απ' όλα, Χαιρετίζουμε ε, το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη βούληση που επέδειξε να ε, υποβάλει δύο πολύ επίκαιρες ε, εκθέσεις εν ώψη και των διαπραγματεύσεων μετά κατά τη διάρκεια και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ήθελα να τονίσω επίση τι θετικέ εξελίξει που δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο βαθμό συνένεση και σύγκληση μεταξύ των δύο εκθέσεων. και σύγκλησή του με τα όσα παρουσίασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Λευκή Βίβλο και το ε, έγγραφο για το μέλλον των ευρωπαϊκών δημοσίων οικονομικών. Και σίγουρα και τα όσα προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να ανεβάσουν τον προπολογισμό στο 1,3 του ΑΕΕ ε των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει βέβαια ότι σίγουρα υπάρχει σημαντική πίεση προς τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να αντιμετωπίσει και να καλύψει όλες τις ανάγκες και προκλήσεις και να πετύχει όλους τους στόχους που έχουν ε, τεθεί σε πολιτικό επίπεδο. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή την κοινή βούληση να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις εν γέρος πριν από τις ε, ευρωεκλογέ του χρόνου για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί και γιατί ξέρουμε ότι η εναλλακτική δεν είναι και τόσο θετική. Είναι θετικό ε, το γεγονός ότι περίπου θα συμπέσουν όλα αυτά με την ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και οι εναπομείναντες 27 θα μπορούν να δείξουν μια κοινή συλλογική πρόταση ε, που θα θεσπίζει κοινού στόχους και τους πόρους που θα πρέπει να διατεθούν για την επιτευξή τους. Για τους ιδίους πόρους, Και πάλι υπάρχει ευρεία συνένεση και σύγκληση μεταξύ των όσων αναφέρατε εδώ σήμερα και των όσων έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Reflection Paper. ενδεχομένως να μην ε, συμπίπτουμε ακριβώς ε, στις προτάσεις, στις ε, συγκεκριμένες προτάσεις για τους επιμέρους πόρους ή φόρους, αλλά γενικά το επίπεδο φιλοδοξίας και το σκεπτικό είναι το ίδιο. Και σίγουρα συμφωνούμε ότι απαιτείται μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, που είναι αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού πακέτου. Εκφράζω λοιπόν την επιθυμία αυτή η διαδικασία, αυτός ο ανοιχτός διάλογος που έχει ξεκινήσει το τελευταίο χρόνο και ο Επίτροπος Σέτιγκερ ε, συμμετέχει στην διαδικασία σε πολλά επίπεδα, ατύπως και επισήμως. προκειμένου με όλο αυτό το προπαρασκευαστικό έργο να ανοίξει ο δρόμος για μια αποτελεσματική διαδικασία διαπραγματεύσεων μέσα στο επόμενο έτος περίπου για να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό εγκαίρως πριν από τις ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέζα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το σημείωμα που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 14 Φεβρουαρίου με ε, ακριβώς εν ώψη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 είναι εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον γιατί ε, μας δίνει ορισμένες ε, μεταβλητές που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στο επόμενο ΠΔΠ. Καλό λοιπόν τους δύο συνεισηγητές να πάρουν το λόγο συμπερασματικά. Ξεκινούμε από τους συζητητές για τους ιδίους επόρους. Α, έχει γίνει αυτό ήδη. Λοιπόν, οι εισηγητέ για του ιδίου πόρου έχουν ήδη πάρει το λόγο συμπερασματικά. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Όλμπριχτ. Ευχαριστώ. Σίγουρα υπάρχουν και ορισμένα δύσκολα ζητήματα, όπως το θέμα της ευελιξίας, διατήρησης ε, των ε, πιστώσουν που δεν έχουν δαπανηθεί. Γιατί έχουμε διαφορετικά όρια και κατόφλια για τους μηχανισμούς ευελιξίας και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, αυτό δεν δημιούργησε όμως μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό επικεντρωθήκαμε στα άλλα πιο ακαθόδη ζητήματα. Όμως, κατά τη συζήτηση αυτή για το ΠΔΠ θα ήθελα να επισημάνω ότι παρατηρούμε και το τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, βλέπουμε τη θέση επιμέρους κρατών μελών, όπως προκύπτει μέρα με τη μέρα. Και είχαμε αρκετές συναντήσεις με πρέσβεις ε, των κρατών μελών που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερως η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι σημαντικό να το επισημάνουμε ενδιαφέρεται κατά τη μέλη τι κάνει το Κοινοβούλιο, γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει θέση. Να επισημάνω εδώ τη θέση της γερμανικής ή της γαλλικής κυβέρνησης ή της ιταλικής κυβέρνησης ε, που ακούσαμε σήμερα. Και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα γύρω από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και μας βοηθάει να καταλάβουμε τη δυναμική ε, εντός του Κοινοβουλίου. Και αυτό συνδέεται και με τι διαπραγματεύσει στη Γερμανία κτλ. Παρατηρούμε λοιπόν τι εξελίξει και θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για τα επιχειρήματα που θα ανακύψουν. Δεύτερο, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουμε αναπτύξει ε, στο κείμενο, ξέρουμε όμω ότι είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν θέλουμε να αντιδράσουμε σε κάτι το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Για συγκεκριμένα έργα ή ιδέες. Για παράδειγμα, στη δέσμη για την Ευρωζώνη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Ξέρουμε ορισμένα στοιχεία, αλλά το ποιος θα, θα το πληρώσει, ποιος θα συμμετάσχει, τι ακριβώς θα περιλαμβάνεται, δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Γι' αυτό και δεν αναπτύσσουμε αυτό το σκέλος. Δεύτερον, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα ταμεία συνοχής. Ε, στην πολιτική συνοχή. Ξέρουμε ότι γίνεται μια εσωτερική συζήτηση στην Κομισιόν να διαχωρίσει το ESF από τη συνοχή. Αλλά δεν μιλάμε γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και αν είναι να γίνει, που εγώ το απέφχομαι, θα αλλάξει τελείως η συζήτηση για την πολιτική συνοχή. Τρίτον, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το ενιαίο Ταμείο Επενδύσεων. Γίνονται κάποιες προκατακτικές παρατηρήσεις, όμως ξέρουμε ότι γίνεται και πάλι έντονη εσωτερική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν νομίζουμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε αυτή τη στιγμή ε, χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε να το κάνει αυτό μέχρι το Μάιο. Και κάτι τελευταίο. Μετά ε, το paper της περασμένης εβδομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχω περιέλθει σε μια σύγχυση, γιατί αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τα όσα μα παρουσίασε η Επιτροπή του τελευταίου μήνε. Πολύ διαφορετικό το περιεχόμενο. Πρέπει να δούμε ποιο από τα δύο ισχύει. Αυτό που μας έδειξε, που μας παρουσίασε ε, ο Επίτροπος Έτιγκερ ή αυτά που βρίσκουμε στο paper. Ίσως το paper είναι μια πρόκληση προς ε, το Κοινοβούλιο αλλά όταν λένε ότι θέλουμε να μειώσουμε ε, κατά 10% τη συνοχή και τα γεωργικά, αλλά στο paper ε, λένε να γίνει περικοπή 15% ή 30%. Αυτό διαφέρει πολύ από το 10% που ακούσαμε στη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Οπότε, ποιες είναι οι προθέσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική μας θέση είναι σαφής. Δεν ζητούμε κάτι από το Συμβούλιο. Λέμε, αυτή είναι η δική μας θέση, τελεία, 1,3. Εμείς περιμένουμε τις απαντήσεις της ε, Επιτροπής. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό το έγγραφο πραγματικά είναι προκλητικό και το θεωρώ εξαιρετικό γιατί ε, θέτει τους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων ενώπιον των ευθυνών τους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε μια σειρά πράγματα και να μην αλλάζουμε τίποτα στον προπολογισμό. Οπότε αναδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο τις αντιφάσεις μεταξύ λόγων και έργων. Κύριε Τωμά. Ναι. Κοιτάξτε, με ενοχλεί που είχαν κάνει διάφορες ερωτήσεις ε, και τώρα έχουν φύγει, αλλά θα επιχειρήσω παρόλα αυτά να απαντήσω. Ιδιαίτερα στα δικά σας ε, ερωτήματα κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς γι' αυτό αρχίζω με εσάς, γιατί εσείς είστε εδώ. Ε, γι' αυτό που είπε ο κύριος Ντεπρέ για την διάρκεια και τη δημοκρατία, δηλαδή για την πενταετή περίοδο του ΠΔΠ. Καταρχάς, ε, υπάρχουν ε, ε, τα όνειρά μας και μετά η πραγματικότητα. Αυτό που θα θέλαμε, το δανεικό, θα ήταν 5 ε, συν 5. Αλλά αυτό δημιουργεί προβλήματα για, το δεύτερο, για τη δεύτερη πενταετή περίοδο. Δηλαδή θα δημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα πριν από τις επόμενες εκλογές. Άρα υπάρχει αυτό το θέμα. Δεύτερον, στα πλαίσια του ΠΔΠ, του τωρινού, υπάρχει η υποχρέωση η Κομισιόν να υποβάλει τις προτάσεις της πριν τις 31 12 17. Και τελικά δεν τη σεβάστηκε αυτή την προθεσμία γιατί θα κάνει τις προτάσεις της ε, το Μάη του 18. Αλλά τα είχαμε προβλέψει όλα αυτά. Αν διαβάσετε τις συμβαστικές προτάσεις για την παράγραφο 20 και την παράγραφο 21, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο της ευελιξίας, αλλά και των αρμοδιοτήτων κάθε κοινοβουλίου για τον προπολογισμό, προβλέπεται μια υποχρεωτική αναθεώρηση. Όχι μια αναθεώρηση όπως προβλεπόταν για το τελευταίο πλαίσιο. Δεν ξέρω να θυμάστε. Είχαμε όλες αυτές τις ε, ε, λεξιλογικές συζητήσεις αν θα είναι review, ε, αν θα είναι revision θέλαμε να έχει, υπάρχει δυνατότητα το Κοινοβούλιο να προτείνει τέτοια αναθεώρηση. Αλλά έπρεπε να συζητήσουμε ακόμη και τους όρους. Τώρα το κείμενό, το κείμενό μας είναι σαφέστατο. Προβλέπεται υποχρεωτική αναθεώρηση. Δηλαδή, όχι μόνο κατά τη διάρκεια κάθε θητείας, δηλαδή κάθε κοινοβούλιο, θα ψηφίσει είτε το ΠΔΠ, είτε την αναθεώρησή του, αυτός είναι ο συμβιβασμός της παραγράφου 20, και για το επόμενο κοινοβούλιο, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, μέσω της συμβαστικής διατύπωσης παραγράφου 21 είναι υποχρεωτικό να υπάρξει κατά τη διάρκεια της θητείας υποχρεωτική αναθεώρηση. Αυτά λοιπόν τα προβλέψαμε. Και εγώ θα προτιμούσα. Είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, όπως και άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα των συμβαστικών ε, διατυπώσεων. Και εγώ θα ήθελα κάθε πέντε χρόνια. Αλλά ορισμένοι είπαν ότι Υπάρχουν θέματα πολιτικής και εσείς ε, που ήσασταν και παλιά πρόεδρος ε, νομαρχιακού συμβουλίου. Υπάρχουν ε, οι ευρωπαϊκές διαδικασίες και μετά υπάρχει η διαδικασία εφαρμογής των αποφασιστέντων από τα κράτη-μέλη. Και ορισμένη πολιτικοί μπορεί να είναι πιο ευέλικτη, αλλά άλλοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η συμβαστική πρόταση 5 5 με υποχρεωτική λοιπόν αναθεώρηση κάθε 5 χρόνια κάτι που δίνει de jure και όχι de facto μια πολύ σημαντική ευελιξία, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα. Ε, τώρα, ο κύριος Σόλε έφυγε, αλλά να απαντήσω. Για την ε, κοινή γεωργική πολιτική, όπως είπε και ο κύριος Όλμπριχτ, δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Προϋπολογισμών να ρυθμίσει τα θέματα περιεχομένου. Και δεν είναι μέσον μέσω του ΠΔΠ που θα αποφασίσουμε το περιεχόμενο των προγραμμάτων. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να διατηρήσουμε τις συνολικές χρηματοδοτήσεις. Γιατί αναφέρθηκε στην ΚΓΠ. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν αυτή τη συμβαστική διατύπωση υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να διατηρηθεί όχι μόνο η χρηματοδότηση αλλά και το περιεχόμενο της γεωργικής πολιτικής, άλλοι θέλουν να την αλλάξουν, αλλά παρόλα αυτά θεωρούν ότι πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοδότησή της. Εμείς απλώς ασχολούμεθα με την δημοσιονομική πλευρά του θέματος. Δεν συζητάμε την ουσία. Δεν συζητάμε τη συζήτηση για τις νομικέ βάσεις. Αυτό θα προκύψει κατόπιν. Αφού καθοριστεί το πι δελτα πι. Λοιπόν, για πολλά θέματα θεωρήσαμε ότι δεν έχει ένα να εισέλθουμε στο περιεχόμενο των πολιτικών. Δεν είναι δικό μας θέμα, δεν πρέπει να συζητηθεί από αυτήν οι παρόμοιες μελλοντικέ εκθέσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Όλμπριχτ και Τομά για αυτές τις τελικές σας ε, διευκρινήσεις. Να μην επαναλάβω, αλλά ε, να πω παρόλα αυτά Εάν οι εκλογές του 19 προκαλέσουν ε, νέες επιθυμίες πολιτικών και το ΠΔΠ είναι το ελάχιστο πλαίσιο, τότε θα πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα αμέσως μετά τις ε, εκλογές της επόμενης χρονιάς. Ούτως ώστε να αυξηθεί αν χρειάζεται ο ενωσιακός προϋπολογισμός, ιδιαίτερα εάν επιτύχουμε να μειωθούν οι εθνικές συνεισφορές. Η Δευτέρα Μαΐου είναι η επόμενη σημαντική ημερομηνία για μας γιατί ο Επίτροπος μας είπε ότι τότε θα υποβάλει τις προτάσεις της για το επόμενο πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να περάσουμε τώρα στην παρακολούθηση της ομάδας για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Θα συζητηθεί και κλεισμένο των θυρών μία σύντομη διακοπή για να αποχωρήσουν όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν.